το εξέλιξη έργο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ νομίζω ότι θα μα διαφωτίσουν καλύτερα για το τι είναι το τοπικό σου παραγόμενα τρόφιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και ακολουθεί ε, η δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα. Θα λάβει πρώτα το λόγο ο κύριος Προεδρεύων. Μπρότσκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανεί το γεγονό ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση όσον αφορά τη μετανάστευση και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε στι προσπάθειέ τη προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί κατάλληλα τη μετανάστευση. Στο Συμβούλιο επανειλημμένως συζητήθηκε η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δράσης της Ελλάδος ε, για το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς επίσης και για τους συνοριακούς ελέγχους. Η πιο πρόσφατη συζήτηση ήταν στις 8 Μαρτίου στο Συμβούλιο ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και τότε ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελλάδα ε, διαπίστωσαν ότι υπάρχει κάποια ε, πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των αιτήσεων ασύλου και τη διεκπαιρέωσή τους. Αλλά ε, σαφώς υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις, κυρίως διότι πρέπει να διασφαλίσουμε αρκετό προσωπικό για τη διεκπαιρέωση των αιτήσεων, αλλά και γιατί πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα κέντρα υποδοχής όλοι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί το Εθνικό Πρόγραμμα Δράση τη Ελλάδο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει και μεγάλη προσπάθεια από πλευρά ε, τη ίδια τη χώρα ε, και θα πρέπει ε, να εφαρμόσει κατάλληλα και να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες όπως ο Frontex και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου αλλά και τα κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Η υπατερμοστία για τους πρόσφυγες επίσης θα μπορέσει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση, εμπειρογνωμοσύνη αλλά και άλλοι διαθέσιμοι πόροι. Τα νέα λοιπόν ότι ετοιμάζεται ένα νέο κέντρο υποδοχή μεταναστών στην περιοχή του Εύρου είναι καθόλου ευπρόσδεκτα σε αυτή τη συγκυρία. Ε, Εντό ολίγου θα λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για το θέμα τη μετανάστευση τη Ελλάδο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τονίσω εδώ το γεγονό ότι εμεί στο Συμβούλιο συζητήσαμε πώ μπορούμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα ε, Προ τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις ε, λόγω της ε, ροή τη μετανάστευση. Εγκρίθηκαν συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο, για ένα πλαίσιο αλληλεγγύης ε, για τα συστήματα ασύλου στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις λόγω των μεγάλων μεταναστευτικών ροών. Και σε αυτό το πλαίσιο αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό αυτό ο μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση που περιέχεται στο κανονισμό Δουβλίνο 2. Ο κανονισμό αυτό ε, περιλαμβάνεται και στο σχέδιο τροποποίησης που έχουμε για το Δουβλίνο 2 και προωθήσαμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξεκινήσουν τριμερείς συζητήσεις επί του ζητήματος. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί εφαλτήριο το οποίο θα μας επιτρέψει να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις όπως αυτή την οποία διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Επιπλέον, έχουμε στη διάθεσή μας και μια εργαλειοθήκη η οποία θα μας βοηθήσει να συνδράμουμε χώρες οι οποίες ε, μπορεί να έχουν ανάγκη βοήθειας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία σε επίπεδο Σέγγεν και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και επίσης το Συμβούλιο συμφωνεί ότι ο ρόλος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να υπάρξει ε, προαγωγή της συνεργασίας με τρίτες χώρες και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με αποτελεσματικό τρόπο και να διαβιβαστούν καταλήλω. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ε, μέσω πρακτικής συνεργασίας. Έτσι θα ενισχυθεί η αλληλεγγύη. Θεωρούμε ότι η αλληλεγγύη είναι μια πολύ σημαντική αρχή και αυτό θα πρέπει να εκπεφραστεί και με πρακτική και απτή συνεργασία. Ως ακρογωνία ολίθο λοιπόν έχουμε την αλληλεγγύη και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης τη Ελλάδο. Το Συμβούλιο υποστηρίζει την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης και επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι επέλεξε να συζητήσει το θέμα αυτό σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση του, Ευρωπαϊκού, του ελληνικού συστήματο μετανάστευση και ασύλου μαζί με του κατάλληλου ελέγχου στα σύνορα δεν είναι ευζωτική σημασία μόνο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για του ίδιου του μετανάστε, του ετούντε άσυλο και του πρόσφυγε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την Επίτροπο Μάλστρομ να πάρει το λόγο. Αξιότιμοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουμε πάλι να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τη διαχείριση τη μετανάστευση, κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και αυτό συνδέεται και με τι συζητήσει που γίνονται για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, αλλά και αφορά και θεμελιώδη δικαιώματα ατόμων και προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχώ υποστηρίζει τι προσπάθειε τη Ελλάδα να αναμορφώσει τι πολιτικέ ασύλου και μετανάστευση. Ε, κατήρτισε ένα πρόγραμμα δράση, όπω είπε και ο Υπουργό, για το άσυλο και τη μετανάστευση και έχει γίνει πρόοδο σε κάποιους τομείς. Δύο νέες υπηρεσίες ιδρύθηκαν, ένα, ε, μία για την εξέταση ε, των αιτήσεων και μία άλλη για την αρχική υποδοχή. Είναι σημαντικό. Πέρσι το ΙΑΣΟ, το ε, Γραφείο Ασύλου έστειλε υποστήριξη και ε, παροχή συμβουλών με υπηρεσίες στην περιοχή του Εύρου που είναι η πιο προβληματική περιοχή. Αυτές οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν φέτος και θα ενταθούν έτη περαιτέρω. Επίσης ε, έχουμε και τεχνική υποστήριξη με αποστολές στην Task Force για την Ελλάδα, με ε, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στη Frontex, την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για μια συνολική προσέγγιση. Εξακολουθούμε να καταβάλουμε προσπάθειες ε, για να συμμετέχουν περισσότερο οι τουρκικές αρχές και να αποτρέπουν τη διαβίβαση και τη διαμετακόμιση μέσω της τουρκικής επικράτειας. Θα πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Εύρο είναι είναι Οι συνθήκες ε, ε, όπου ε, κρατούνται ή διαβιούν οι ετούντες άσυλο και οι μετανάστες είναι προβληματικές. Χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες από τις ελληνικές αρχές για μηχανισμούς έγκαιρης βοήθειας και ανακούφισης προς εκείνους που περνούν τα σύνορα θα πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα προσωρινής υποδοχής ε, για ε, ευάλωτες ομάδες ε, και κάποια θέματα ασφαλείας στην περιοχή. Επανειλημμένα έθεσε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ελληνικών Αρχών ότι μπορεί η μη συμμόρφωση και συνέχεια να οδηγήσει και σε νομικές επιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και πολλά όργανα στα κράτη-μέλη, αλλά η ίδια η Ελλάδα οφείλει να δρά ε, συμμορφούμενη προς το διεθνές δίκαιο αλλά και το κοινωτικό. Ε, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε στρατηγική και τακτική υποστήριξη στην Ελλάδα για αναμόρφωση του συστήματος. Αυτό σημαίνει και επιπλέον χρηματοδότηση ε, και επιμελητία αλλά και πραγματογνωμοσύνη επιτόπου, συνεργασία με τις εθνικές αρχές, οργανισμούς, ε, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ε, και την ύπατη αρμοστία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρηματοδοτεί γενναία την Ελλάδα 309 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα απορρόφησης από την ελληνική πλευρά. Ε, και πολύ λίγα από τα κονδύλια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί. Για τις άμεσες ανάγκες πρόσφατα ε, δώσαμε και ένα ποσό ε, από το Ταμείο Προσφύγων 3,75 εκατομμύρια ευρώ για τις πιο επίγουσες ανάγκες και θα πρέπει να απορροφηθούν αυτά. Είναι σημαντικό ο μηχανισμός να ε, εξομαλυνθεί σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση των κονδυλίων. Η ε, υποστήριξη δίνει και η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη απορρόφηση και να προωθηθεί το πακέτο της μεταρρύθμισης. Το Δεκέμβριο εμπειρογνώμονες ε, καταστάθηκαν στην Αθήνα για να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να απορροφήσει αυτά τα κονδύλια. Πρόταση αναδιατύπωσης επίσης για τον κανονισμό του Δουβλίνου όπως και το υπόλοιπο ε, πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και την προστασία των ετούντων άσυλων προσβλέπω ε, στην Προεδρία για να ε, βεβαιωθεί ότι θα αρχίσει ο τριμερής διάλογος για αυτά τα θέματα και για άλλα συναφή και σχετικά με το πακέτο ασύλου. Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια στιβαρή και γερή πολιτική ασύλου. Να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη να είναι σημαντικό ε, το θέμα της διεθνούς προστασίας ε, εκείνων που την έχουν ανάγκη. Είναι κοινό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και εδώ και καιρό. Χρειάζονται κοινοί κανόνε και μεγαλύτερη ελεγγύη και η ανάγκη αυτή είναι όλο και πιο πιεστική. Υψηλά πρότυπα, μεγαλύτερη συνεργασία έτσι ώστε οι άσυλο να έχουν ίση μεταχείριση όπου και αν την αίτηση και όσοι χρειάζονται χρειάζονται προστασία να έχουν πρόσβαση στην προστασία. Ένα δίκαιο σύστημα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ε, επιμεριστούν τις ευθύνε γι' αυτό. Το σύστημα του Δουβλίνου χρειάζεται να συμπληρωθεί, ε, να αντιμετωπίσει το κακό στη ρίζα του, ε, τα προβλήματα, τα ελλείμματα και λήψεις να αντιμετωπιστούν χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση γιατί τίθεται και θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμετέχουμε, θα εξακολουθήσουμε, συμμετέχουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εκτιμώ και την ισχυρή δέσμευση του Συμβουλίου και άλλων οργανισμών, αλλά την κύρια ευθύνη βεβαίως φέρει ε, η Ελλάδα και οι ελληνικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Μάλστρομ. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές και τις ομιλήτριε εξ των πολιτικών ομάδων. Και ήθελα πρώτα να παρακαλέσω την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να πάρει το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χωρίς αμφιβολία, είναι προτιμότερο <clears throat> να προλαμβάνει κανείς παρά να θεραπεύει. Συμφωνώ απολύτως με την Επίτροπο σε όσα είπε για τα ατομικά δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν όσοι αιτούνται άσυλο εκείνο που δεν σημείωσε ε, και δεν έκανε σαφές στο ακροατήριο είναι ο τεράστιος αριθμός αυτών που μπαίνουν στην ελλάδα ως παράνομοι μετανάστες. όταν η τουρκία έχει έχει απελευθερώσει τη βίζα για όλες τις χώρες της περιοχής και της μεσογείου και με 50 ευρώ μπορεί κάποιος από την τρίπολη της λιβύης να έρθει στην ισταμπούλ και εν συνεχεία να έρθει οδικός στα σύνορα με την ελλάδα αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται. αυτοί που μπαίνουν εκεί τους οποίους φέρνουν οι διάφοροι έμποροι στην κυριολεξία έμποροι ανθρώπων δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η καταγωγή τους ούτε ποια γλώσσα μιλούν δεν έρχονται με χαρτιά και βεβαίως ζητούν όλοι άσυλο. όταν λοιπόν μπαίνουν 300 ή 500 άνθρωποι την ημέρα από τα σύνορα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς ένα τόσο πολύ μεγάλο αριθμό. γι' αυτό και συμφωνώ με την επίτροπο ότι χρειάζεται διαφοροποίηση στο δουβλίνο 2 κυρία Μέλστρομ και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαπιστώνετε και θέλετε να το ενισχύσετε. Όταν η Ελλάδα λοιπόν φέρει συνολικά το 90% του βάρους της πίεσης της παράνομης μετανάστευσης αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση να γίνουν πάρα πολλά κέντρα στα οποία θα κρατηθούν υπό ανθρώπινες συνθήκες οι μετανάστες και θα γίνει μια προσπάθεια να επαναπροωθηθούν αλλά η λύση του προβλήματος είναι μία κυρία επίτροπε να υποχρεωθεί η τουρκία να εφαρμόσει τη σύμβαση που έχει με την ευρωπαϊκή ένωση για την επαναπροώθηση και να υποχρεωθεί να εφαρμόσει και τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την ελλάδα από το νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια υποψήφια χώρα η οποία θέλει να αναγνωρίζει ή να μην αναγνωρίζει τις συμφωνίες με την ευρώπη στα δικά της μέτρα. οφείλει να υποχρεωθεί η τουρκία να εμποδίσει αυτή την τεράστια πίεση. κατά τα άλλα κανείς στην ελλάδα δεν θέλει να στερήσει ανθρώπινα δικαιώματα από τους ανθρώπους αυτούς. μετέχουμε πλήρως στην ένωση και στις αντιλήψεις και στις αξίες που υπερασπιζόμεθα κυρία επίτροπε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να υπερασπισόμεθα. αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά ουσιαστική στήριξη από την ένωση το συμβούλιο το κοινοβούλιο και εσάς βεβαίω που σωστά διαχειρίζεστε την υπόθεση αυτή. Σας Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γεννάκου. Ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κυρία Γκυγιόμ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ η ανησυχία που προκαλεί η κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα δεν είναι κάτι καινούριο. Χρειάζονται σημαντικά μέτρα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη έχουν ληφθεί κάποια για να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στι ανάγκε. Σήμερα βλέπουμε ότι είναι οξύτατο το πρόβλημα και ένα προεδρικό διάταγμα το 2010 υλοποιείται στην Ελλάδα που λέει ότι θα πρέπει να συγκεντρώνονται οι λαθρομετανάστε και οι αιτούντε άσυλο, ιδίω όσοι είναι υποπτοί ότι μπορεί να είναι φορεί ε, μεταδοτικών ασθενειών. Τέτοια μέτρα θα ήταν βεβαίω πολύ ανησυχητικά, εφόσον υλοποιούνται, για πολλού λόγου. Πρώτα απ' όλα, επειδή του πλέον ευάλωτου μπορεί να του θεωρούν υπόπτου ε, και αυτό αποτελεί περίπτωση διακριτική μεταχείριση. Επίση, γιατί είναι πολύ επισφαλή κατάσταση των μεταναστών και των μεταναστών στην Ελλάδα. Και βεβαίω το θέμα είναι πώ ε, γίνεται ποιε είναι οι συνθήκε κράτηση των ελευθερομεταναστών στην Ελλάδα. Ε, άτομα τα οποία μπορεί να χρήζουν διεθνού προστασία. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το θέμα να ενσκύψουμε πόσο μπορεί να είναι η πραγματικότητα αυτή. Θα πρέπει επίση να δούμε και άλλα ζητήματα που συνδέονται με αυτό, διότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ε, εξακολούθηση αυτή τη συζήτηση που θα πρέπει να είναι πολύ συνετή και ε, σε συνθήκε ψυχραιμία, ώστε να βρούμε συγκεκριμένε λύσει. Υπάρχει και πρόβλημα χρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ρωτήσω τι δράσει ε, έχουν αναλυφθεί πρώτε και ε, σε αυτή την περίοδο και τι προβλέπετε για το μέλλον και να μας πείτε πώς λόγω χάρη πραγματοποιείται η ταυτοποίηση των ατόμων που χρήζουν διεθνού προστασίας και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ανάλογη διαδικασία, πώς εξετάζονται οι αιτήσει τους και οι αιτήσει εισόδου γιατί μας, είπε, μας είπαν, ε, ακούσαμε ότι η Ελλάδα επαναπροωθεί κάποιες φορές τέτοια άτομα αλλά σίγουρα οι προσπάθειε να ενισχυθεί αυτό το κράτο μέλο σε τεράστιε μεταναστευτικέ πιέσει θα πρέπει να ενισχυθούν. Αλλά και το διεθνέ δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να υπερισχύουν σε συνθήκε αμοιβέ εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών. Το όνομα τη ομάδα των φιλελευθέρων, η κυρία Γκρίσμπεκ, παρακαλώ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλήσαμε για προκλήσεις Πράγματι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση τεραστίων διαστάσεων για την Ελλάδα. Όμω είναι μια πρόκληση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε κάποια απόκριση για την εικόνα μα παγκοσμίω και βεβαίω στα μάτια των πολιτών. Θα μπορούσε κανεί να φανταστεί ότι με το τέλος του 20ου αιώνα την πτώση του τείχους του Βερολίνου θα περνάγαμε σε... δεν θα περνάγαμε στην ε, δημιουργία νέων τυχών στην περιοχή της Ευρώπης. Κι όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα φαίνεται να επιδιώκει κάτι ανάλογο. Για να αντιμετωπίσει μια τέτοια πραγματικότητα, πιεστική πραγματικότητα, όπως είπε η συνάδελφος Γιαννάκου, 300 άτομα ημερησίως από γειτονική χώρα, χώρα διέλευση, στην Τουρκία. Αλλά όχι από πολίτε τη χώρα αυτή, από πολλέ άλλε χώρε του υπόλοιπου κόσμου. Θα ελπίζαμε να μην επανελευθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και βεβαίως εδώ δημιουργούνται ανθρωπιστικές συνθήκες απαράδεκτες. Ε, μιλάμε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανθρώπινα δικαιώματα που διαρκώ ε, επιδιώκουμε να προστατεύουμε, να διασφαλίζουμε ως το πολυτιμότερο αγαθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε και γέννησε. Εδώ λοιπόν τα μηνύματα είναι σίγουρα πολλά και αλληλένδετα. Αλλά δεν θα πρέπει να πούμε στι τεχνικέ λεπτομέρειε. Να σταθούμε στο ότι η αλληλεγγύη, όπω την παρουσίασε η κυρία Μάλστρομ μέσω τη κοινή ευθύνη μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών χρηματοδότηση είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί. Χρειάζεται δε κονδυλίων ευρωπαϊκή προέλευση ώστε να δοθεί αποτελεσματική πρακτική βοήθεια και να αποκριθούμε με τρόπο ε, σύμφωνο με τα δικαιώματα του ανθρώπου ε, και τις ε, ανάλογες ανάγκες στην προστασία αυτών των ατόμων. Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε ότι η συζήτηση αυτή έχει φουντώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι χρειαζόμαστε κείμενα, ένα, ένα σύστημα δικαίου το οποίο να επιτρέπει την πραγματική αλληλεγγύη, την χειροπιαστή αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και για τα ελληνικά σύνορα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε το πλωστάσιο κειμένων που διαθέτουμε να αξιοποιηθεί. Και δεν θα πρέπει να σφάλουμε στα πλαίσια τη συζήτηση, διότι στη Γαλλία μιλάμε για προστασία των εσωτερικών μα σύνορων, των γαλλικών σύνορων. Όχι, εδώ μα ενδιαφέρουν και τα εξωτερικά μα σύνορα, στα πλαίσια του ανθρωπισμού που μα διέπει. Επίση, Πρόεδρε, το τρίτο μήνυμα που φαίνεται να υπερισχύει μέσα από τα λεγόμενά μα λεγόμενά μα είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση να δημιουργηθεί ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου. Να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αναπτυξιακή βοήθεια και τι εταιρικέ σχέσει με τι χώρε του Νότου, ώστε οι πολίτε των χωρών αυτών να μην επιδιώκουν να έρθουν στο Ελντοράντο που δεν είναι Ελντοράντο. Ευχαριστώ γαλάζια κάρτα, κυρία Γκρισπέκ, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Δέχεστε, παρακαλώ. Σε σχέση με τα σχόλια της ε, εξαίρετη συναδέλφου για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, πέρυσι στην Λαμπεντούζα κατέφθασαν περίπου 60.000 συνολικά υπήκοοι τρίτων χωρών από τη Βόρειο Αφρική μετά από τις όλες ε, εξελίξεις που είχαμε στην περιοχή. Στην Ελλάδα, κυρία συνάδελφε, φτάνουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 120.000 υπήκοοι τρίτων χωρών στα ελληνικά σύνορα με βάση μόνο τι συλλήψει και τα στοιχεία τη frontex. πιστεύετε πραγματικά ότι η ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει μόνη τη να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση τη στιγμή μάλιστα που έχει έξι φορέ μικρότερο πληθυσμό από την ιταλία. Ευχαριστώ, ε, κυρία euh, ναι, ευχαριστώ. Βρίσκεστε στο πίσω μέρο τη αίθουσας. Βεβαίω έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα τη δυσκολία τη Ελλάδα να ανταποκριθεί μόνο τη σε τέτοιε ανάγκε. Βεβαίω, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη Σάμο. Όμω είδαμε την κατάσταση επικράτη στην Ελλάδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πήγα και στη Λαπεντούζα, όπω λέτε, και είδα πραγματικά πόσο πολύ τα προβλήματα είναι εκτεταμένα. Όμω, θα πρέπει εφαρμόζοντα την αλληλεγγύη στηρίζοντα την Ελλάδα που είναι και μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναζητήσουμε τι κατάλληλε απαντήσει. Επί τη ουσία, θα πρέπει όλε οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθούν στην υπηρεσία αυτή του στόχου. Καταλαβαίνω τι ίδιε δυσκολίε τη Ελλάδα. Εδώ αισθάνομαι Ελληνίδα και εγώ μαζί σα. Ευχαριστώ κυρία Κυρία Φλότρο, παρακαλώ. Εξ ονόματος για πόση ώρα παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα, ε, τα ΔΕΚ, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες οργανώσεις έχουν κρούσει τον κρόδωνα του κινδύνου που τον άκουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκτοτε η Ελλάδα έχει ένα εθνικό σχέδιο για το άσυλο και τη μετανάστευση, αλλά θα πρέπει να ε, καταλάβουμε σήμερα ότι στα κέντρα κράτησης η κατάσταση και έχω ε, επισκεφθεί είναι ύβρις προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και από την αρχή του χρόνου έχουν χάσει τη ζωή τους πολύ προσπαθώντας να διασχίσουν τον Εύρο οι μη κυβερνητικέ οργανώσει σήμερα με την οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα διαπιστώνουν την ακραία αύξηση ρατσιστικών επιθέσεων και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Έχουμε 63 περιπτώσεις, εκ των οποίων 18 από την αστυνομία στο τελευταίο εξάμεινο του 2011. Και είναι σαφές ότι σε μια προεκλογική περίοδο σήμερα στην Ελλάδα ακούμε ε, προτάσεις ε, εξωφρενικές ε, και μια κούρσα ιδιαίτερα ξενόφοβη και κατά των μεταναστών. Κατασκευάζονται κέντρα κράτησης, αλλά κυρίως η πρόταση αυτή ε, στοχεύει στη στάθμευση ε, των μεταναστών και των άσυλο που υποτίθεται ότι είναι ασθενείς. Και μάλιστα πολιτικοί ηθήνοντες χαρακτηρίζουν βόμβα για την ασφάλεια της χώρας το μεταναστευτικό και απέναντι σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαντήσει με τις αξίες της, με τα μέσα της και με τις αρχές της συνεργασίας και αλληλεγγύης. Και θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη, αντί να απειλούν την Ελλάδα ότι θα τη διώξουν ε, από το Σέγγεν, που είναι τελείω σκανδαλώδης πρόταση, ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη εκφράζουν ε, ανοιχτά τη θλίψη του στο γεγονό ότι του απαγορεύει το δικαστήριο να στέλνουν στην Ελλάδα ετούντε άσυλο στα πλαίσια του Δουβλίνου 2. Αυτή η υποκρισία είναι αφόρητη ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλη ευθύνη εδώ για να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί τι βασικέ μα θεμελιώδεις αξίε. Επίση πιστεύω ότι και με τη Τουρκία θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ε, για τις συμφωνίες επανεζοχής και επαναπροώθησης. Η Τουρκία ζητάει αμοιβαιότητα. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε να συζητούμε για απελευθέρωση των θεωρήσεων. Η πρόεδρος τελειώνεται, παρακαλώ, τελειώνω. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία δέχεται χιλιάδες ε, πρόσφυγες κάθε μέρα στα σύνορά της με τη Συρία. Θα πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε ένα στο μπαλάκι στον άλλον και να αναλάβουμε με αλληλεγγύη ε, τη βασική μας ε, ευθύνη. Ευχαριστώ. Δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τριανταφυλλίδη από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με τον οποίο και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των ομιλητών και των ομιλητριών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Θέλω να σας πω ότι έχω όλη την καλή διάθεση να είμαι ευέλικτη ως προς το χρόνο γιατί έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας αλλά ε, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα για να υπερβαίνουμε το χρόνο μας σχεδόν κατά ένα ολόκληρο λεπτό. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ κυρία πρόεδρε η κατάσταση των μεταναστών στην ελλάδα φανερώνει πολλά για την γενικότερη κατάσταση πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας καταστολής κατάφορων διακρίσεων εκμετάλλευσης εκφοβισμού είναι μόνο λίγα από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα. μαζικές κρατήσεις μεταναστών σε φρικτές συνθήκες στερούμενοι ακόμη και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και ενίοτε θύματα αστυνομικής βίας και ταπεινωτικής μεταχείριση αλλά και για όσου δεν κρατούνται οι περισσότεροι του ζουν σε συνθήκε κοινωνικού αποκλεισμού χωρί πιθανότητε κοινωνική ένταξη, πέφτουν θύματα βία και ρατσισμού και εκμετάλλευση από κυκλώματα και εργοδότε. εν ώψη των επικείμενων εκλογών ενισχύεται η αδικία και ο παραλογισμό. οι μετανάστε μετατρέπονται από το κράτο σε αποδιοπομπαίοι τράγοι τη κρίση σε αποδέχτες τη γενικευμένη απελπισία και οργή για την εξαθλίωση παρουσιάζονται σαν υγειονομική βόμβα που απειλεί την υγεία και σαν απόλυτη φορή εγκληματικότητα. ενισχύεται η ξενοφοβική ρητορική και πληθαίνουν οι συλλήψεις και οι επιχειρήσεις σκούπα όπως τις αποκαλούν ως αν μιλάμε για σκουπίδια. μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2011 σημειώθηκαν 60 περιστατικά ρατσιστικής βίας στην αθήνα τα οποία έχουν εξαπλωθεί και αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και μάλιστα με συμμετοχή ανηλίκων οι ευθύνε είναι σημαντικέ και από πλευρά κράτου αλλά και ευρωπαϊκή ένωση. ελπίζουμε ότι η αλληλεγγύη στην οποία έκανε αναφορά ο υπουργό προηγουμένω θα πάψει να είναι απλώ ένα σύνθημα αλλά θα μεταφραστεί σε πράξη σε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου η ευρώπη θα έρθει αρρωγό σε χώρε που είτε λόγω γεωγραφία είτε άλλω πω είναι αδύναμε να αντιμετωπίσουν τι ροέ μεταναστών που η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση εξαναγκάζει να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην ευρώπη. μια αλληλεγγύη που θα πρέπει να είναι σφαιρική να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα αλλά και υποστηρικτική τεχνική βοήθεια για εξέταση αιτήσεων και δημιουργία κατάλληλων κέντρων υποδοχή. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αποφασίσει και να αποδείξει το πραγματικό τη πρόσωπο μυσαλλόδοξη και φοβική ή ισότητα και ειρηνική συνύπαρξη ο δεύτερος δρόμος είναι ίσως πιο δύσκολος αλλά αυτόν επιθυμούμε και αυτό πρέπει να διεκδικούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στους ε, άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές και ομιλήτριες και πρώτα θέλω να παρακαλέσω την κυρία Χολμάιερ να πάρει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευθύς εξ αρχής ε, ήθελα να απευθύνω ευχαριστίες το Γραφείο Υποστήριξη για το Άσυλο που στο μεταξύ ε, με τρόπο πολύ αποτελεσματικό βοηθάει σοβαρά την Ελλάδα ε, και είναι και πολύ αποδοτική η εργασία. Ακριβώς αυτό που ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι ε, για να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής ασύλου. Το, Ευρωπα... Πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να δημιουργηθούν και επιπλέον κέντρα υποδοχής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ε, υποστηρίζεται αντίστοιχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πρέπει τουλάχιστον να υποστηρίζεται και μέσω του Γραφείου για την Υποστήριξη του Ασύλου. Ε, θεωρώ σημαντικό και χρήσιμο εδώ στο Κοινοβούλιο να μην περιγράφουμε πάντα τις δυσκολίες μόνο και τις φρικαλαιότητες αλλά και πολύ συγκεκριμένα να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και να μην ε, ε, ζητάμε από την Ελλάδα που αντιμετωπίζει μια ολέθρια οικονομική και δύσκολη κατάσταση σήμερα, θα κάνει όλα από τη μια μέρα στην άλλη, να έχουμε και ένα ρεαλιστικό σχέδιο και ένα γνώμονα για το μέλλον. Γι' αυτό θεωρώ χρήσιμο. Ε, που ε, ε, σταμάτησαν ε, την επαναπρόθεση στην Ελλάδα των προσφύγων κάποιες χώρες. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να αναπτυχθεί συνεργασία με την Τουρκία. Είπε η Επίτροπος ότι κάνουμε τις προσπάθειες αυτές, αλλά θεωρώ ότι να συνδέεται η πολιτική θεωρήσεων των διαβατηρίων με την επαναπροώθηση είναι ιδιαίτερα προβληματικό ζήτημα. Δεν ξέρω, ε, αντιθεωρήσεις διαβατηρίων δεν μπορούμε να επιλέξουμε το ε, γενικότερο πλαίσιο, να ασχοληθούμε περισσότερο και να περιοριστούμε σε φοιτητέ και επιχειρηματίες, ίσως αυτό να ήταν λύση και για τις χώρες που αυτόν τον καιρό έχουν δυσκολίες να απελευθερώσουν τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Και στην επαναπροώθηση νομίζω θα πρέπει να τονίσουμε και την αστυνομική συνεργασία. Διότι περί αυτού πρόκειται ε, καταπολέμηση δουλεμπόρων που στις πλάτες των καημένων των προσφύγων βγάζουν λεφτά. Και ε, ε, δεν θα πρέπει να έχουμε άχρηστη αντιπαράθεση με τη Τουρκία επί της ουσίας. Ελπίζω η Τουρκία να είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε αστυνομική συνεργασία για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χολμάγια. Κύριε Ρούμπικ, σηκώσατε γαλάζια κάρτα. Σωστά. Καλά σας είδα. Κυρία Χολμάιερ, δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Ρούμπικ. Μάλιστα. κύριο Ρούμπικ, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χολμάγερ γιατί ε, τόνισε και τα θετικά στοιχεία. Δηλαδή, γιατί μπλε κάρτα να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να εντάξουμε μετανάστες στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να κοιτάξουμε τα προσόντα, τις δεξιότητες του καθενός και να δούμε τι χρειάζεται η Ευρώπη, ε, τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις και θετικά να αξιολογηθεί και να ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί στην αγορά εργασία. Χρειάζεται δηλαδή μια λεπτομερή ανάλυση για να φροντίσουμε να απορροφήσουμε όσο γίνεται και να εντάξουμε του ανθρώπου αυτού στην Ευρώπη. Ερώτηση ήταν αυτή. <laughs> Ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάγερ. Ναι, όντω πιστεύω και εγώ ότι σε συνεργασία με το Γραφείο για την Υποστήριξη του Άσυλο και τι ελληνικέ αρχέ ε, θα πρέπει να φροντίσουμε πιο γρήγορα να εντοπίζουμε εκείνους που έρχονται και φτάνουν στην Ελλάδα και θα μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς γιατί ε, πρώτον δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γυρίσουν στην πατρίδα τους και δεύτερον μπορεί να έχουν δεξιότητες, προσόντα και δυναμικό που να μας είναι χρήσιμο και να ε, μας βοηθάει αλλά κυρίως πρόκειται για ενίσχυση προς την Ελλάδα για να υπάρξει καν μια καταγραφή και πιο γρήγορη ταυτοποίηση έτσι ώστε να επιταχυθούν οι διαδικασίες αλλά και να επαναπροωθούνται στις πατρίδες τους εκείνοι που δεν έχουν ε, κανένα λόγο να βρίσκονται στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε προσόντα ούτε δεξιότητες και στη χώρα τους θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες αν είχαν μείνει. Θέλω τώρα να παρακαλέσω τον κύριο Δρούτσα να πάρει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την Επίτροπο κυρία Μάλμστρομ προσωπικά για τον τρόπο που στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Και δεν θέλω να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα που λαμβάνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Η κοινωνική ειρήνη στην Ελλάδα τίθεται σε κίνδυνο. Υπάρχει πλέον και θέμα δημόσιας υγείας και επιπλέον είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει σε ένα λαό που βλέπει τους μισθούς και τι συντάξει του να κόβονται δραστικά πω πρέπει να ξοδέψει χρήματα που δεν περισσεύουν για να βοηθήσει έναν ξένο σε εισαγωγικά. ναι είναι πρόβλημα τη Ελλάδα, και σαφώς στο παρελθόν δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και πιστέψτε με για τι εικόνε που βλέπουμε από τον εύρο κανένα Έλληνα δεν είναι περήφανο. αλλά είναι και πρόβλημα σοβαρό πρόβλημα και για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό ευτυχώ συμφωνούμε σήμερα όλοι και επιτρέψτε μου να πω με όλη την ευγνωμοσύνη μου για την βοήθεια που χορηγείται στη χώρα μου ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει κάνει αρκετά προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής και συνολικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που χρειαζόμαστε. πρέπει να είμαστε τολμηροί και απευθύνω έκκληση προς την επιτροπή και το συμβούλιο να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την αλλαγή του δουβλίνου 2 και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αλληλεγγύη στη διαχείριση των προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών. δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε αυτά μόνο επειδή η σημερινή κατάσταση εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων κρατών μελών με κόστος δυσβάσταχτο κόστο για κάποια λίγα κράτη μέλη όπω την ελλάδα. διότι ένα είναι σαφέ, όσο και καλά να διαχειριστεί η ελλάδα του Ευρωπαϊκού πόρου είναι αδύνατο να παρέχει το υψηλό επίπεδο διεθνούς προστασίας που σωστά έχουμε καθιερώσει στην ευρώπη όταν το 90% των μεταναστών που έρχονται στην ευρώπη έρχονται μέσω της ελλάδας. κυρία πρόεδρε επιτρέψτε μου να κλείσω με την εξής επισήμανση η ελλάδα βρίσκεται όπως γνωρίζουμε σε προεκλογική περίοδο. καλός ή κακός αυτή είναι η πραγματικότητα το θέμα της παράνομης μετανάστευσης έχει ήδη γίνει πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης ιδίως από ακραία κόμματα ο λαϊκισμός δυστυχώς περισσεύει κάποιοι παίζουν εύκολα με τις ευαισθησίες και τους φόβους τους δικαιολογημένους φόβους του κόσμου. χρειάζεται λοιπόν από όλους και απευθύνω έκκληση προς όλους να επιδείξουν την απαραίτητη προσοχή και ευαισθησία στο χειρισμό αυτού του θέματος ειδικά αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Δρούτσα, έχει σηκώσει μπλε κάρτα ο κύριος Χρυσόγελος, ο οποίος θα επιθυμούσε να σας ε, απευθύνει μια ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Χρυσόγελε. Κύριε Δρούτσα, επειδή συμμετείχατε και στην κυβέρνηση πριν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, τι ποσοστό έχει απορροφηθεί από τα 309 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε η Επίτροπος στην Ελλάδα για το θέμα των μεταναστών γιατί αναφερθήκατε σε κόστο, το οποίο δεν μπορούν να πληρώσουν οι Έλληνε. αλλά υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι η ελλάδα του έχει εξαντλήσει. Ε, από του πόρου που, διαθε... διατίθεται για εθελοντικό, ε, για εθελοντική, ε, εθελοντικό επαναπροσ... να επιστρέψουν δηλαδή εθελοντικά στη χώρα του. υπάρχουν 3.000 αιτήσει. πόσες από αυτέ έχουν λάβει απάντηση και έχουν διατεθεί υπάρχοντες πόροι και στο τέλο, πόσε από τι αιτήσει για άσυλο έχουν εξεταστεί και έχουν δοθεί σε αιτούντε άσυλο. Που θα Ευχαριστώ ένα κύριε Χρυσόγελε. Παρακαλώ κύριε Δρούτσα. Κύριε Χρυσόγελε θα μου τρέψετε να πω ότι δεν θα μπω σε αυτό το παιχνίδι να μεταφέρουμε αυτό το σημαντικό και σοβαρό θέμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω μια εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται δυστυχώ στην Ελλάδα αυτά τα ερωτήματα θα σας παρακαλούσα να τα απευθύνετε στην κυβέρνηση και στην ευρωπαϊκή επιτροπή η οποία σίγουρα θα σας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. σας ευχαριστώ. Κύριε Δρούτσα, ε, κύριε Χρυσόγελε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Στην Ελλάδα έχει πράγματι ιδιαιτερότητες γιατί η Ελλάδα ήταν χώρα αποστολής και όχι υποδοχής μεταναστών είναι κοντά σε έφλεκτε περιοχέ και έχει μεγάλο μήκο συνόρων που είναι αδύνατο να κλείσουν αεροστεγώ. αλλά μια ανθρωπιστική και οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική μπορεί να υποφελεί και για του έλληνε και για του μετανάστε όπω έχει δείξει εμπειρία στη γερμανία στο βέλγιο στη ηπα και στην αυστραλία. αυτέ οι χώρε θα ήταν ισχυρέ χωρί μετανάστε πρέπει να αναρωτηθούμε. και πολλοί έλληνε ήταν αυτοί που έπαιξαν ρόλο στην δύναμη αυτών των χωρών. χρειάζεται λοιπόν να τερματιστεί η παθητική στάση που οδηγεί σε ξενοφοβία αλλά και να απομονωθούν οι ακραίε φωνέ υπουργών πολιτικών και κομμάτων που εμποδίζουν αντί να επιλύουν το πρόβλημα με προτάσει για μαζικέ απελάσει, φράχτε στα σύνορα στρατόπεδα κράτηση που δεν είναι μόνο επικίνδυνε αλλά και ανεδαφικέ. αποτελούν κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτούν μεγάλη κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλεία και τεράστιο κόστο απελάσει 400.000 ανθρώπων προτείνουν ορισμένοι. υπάρχουν ρεαλιστικέ και βιώσιμε λύσει που πρέπει να προωθηθούν από την ελλάδα με αλληλεγγύη τη ευρώπη γιατί πράγματι το πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό και να αναλάβει η χώρα τι ευθύνε τη. οι νόμιμοι δρόμοι μετανάστευση και η αποτελεσματική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων για 309 εκατομμύρια μίλησε η επίτροπο η δημιουργία κέντρων πρώτη υποδοχή και κέντρων διαχωρισμού αλλά και εθελοντικό επαναπατρισμό ε, θα αποφορτήσουν την πίεση στην Ελλάδα και θα χτυπήσουν τα κυκλώματα παρανομία. ήθελα να πω επίση ότι αν αποδοθεί σωστά το σύστημα ασύλου. Κύριε Χρυσόγελε, ε, έχετε υπερβεί το χρόνο σα και τα μισό λεπτό. Σα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο ε, Πουζούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ε, θεωρώ ότι η Ελλάδα πάσχει από τα συμπτώματα της μετανάστευσης. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι όπως και άλλες χώρες της ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες είναι ε, είναι χώρα διέλευση, δεν είναι χώρα ε, παραμονή. Οι μετανάστες πηγαίνουν στην Ελλάδα, αλλά δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Θέλουν απλώς να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εκεί. κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι τόσο τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδος όσο και ο αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και η Ελλάδα υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως η Μάλτα, η χώρα μου. Έχουμε το παράδειγμα της Λαμπεντούζα. Οι 60.000 άνθρωποι που φτάνουν στη Λαμπεντούζα δεν θέλουν να παραμείνουν στη Λαμπεντούζα και όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο σφάλει σαφώς. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δούμε πώς να αντιμετωπίσουμε το συλλογικό πρόβλημα της Ευρώπης από κοινού. Θεωρώ ότι τα όσα προτείνει το Συμβούλιο για την ε, ε, με, τροποποίηση του κανονισμού Δουβλίνο 2 πόρα απέχει από την ε, λύση του θέματός μας και γι' αυτό θα πρέπει τα όσα είπε το Συμβούλιο για την Αλληλεγγύη, παρά το γεγονό ότι είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να γίνει κάτι περαιτέρω. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι ευρωπαϊκό. Εάν δεν το κατανοήσουμε, δεν θα υπάρξει λύση. Κύριε η κυρία Φαζόν, παρακαλώ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Δεν είναι στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Παπα-Νικολάου. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να πω καταρχά σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν προηγουμένω ότι οι Έλληνε είμαστε λαό φιλόξενο και διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι στεκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μα από όπου και αν εκείνο προέρχεται και σεβόμαστε τα δικαιώματά του. Πρέπει όμω σε σχέση με τι αναφορέ που έγιναν και τι καταγγελίε από συναδέλφου να πω ότι δικαιώματα έχει και η οικογένεια του ανθρώπου για παράδειγμα που πριν από μερικού μήνε δολοφονήθηκε στι 6 ώρα το πρωί όταν πήγαινε την έγκυο γυναίκα του στο μεευτήριο για να γεννήσει από παράνομου μετανάστε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, διάβασα τη χθεσινή επιστολή των υπουργών εσωτερικών τη γαλλία και τη γερμανία με την οποία ζητούν τη δυνατότητα έκτακτη επαναφορά συνοριακών ελέγχων και συχνά αρχηγοί κρατών το προηγούμενο διάστημα αναφέρονται στη μείωση των αριθμών μεταναστών που επιθυμούν να δέχεται η χώρα του. σε σχέση με τι αναφορέ αυτέ επιτρέψτε μου να τονίσω τα εξή όταν στο σπίτι σου δεν θε να μπουν άλλοι παράνομοι επισκέπτε δεν κλείνει ούτε την πόρτα του σαλονιού ούτε την πόρτα τη κουζίνα. κλείνει την εξώπορτα ασφαλίζει την κύρια είσοδο. αυτή είναι η λύση στο ζήτημα τη παράνομη μετανάστευση στην ευρώπη πρέπει να εφαρμόσουμε την απλή λογική που εφαρμόζουμε και στο σπίτι μα. και εδώ σπίτι μα είναι η ευρώπη και κύρια είσοδο στα εξωτερικά σύνορα τη ευρώπη. και αν ρωτήσετε τη frontex και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία θα σα πούνε ότι η κύρια πύλη εισόδου των παράνομων μεταναστών στην ευρώπη αναφέρθηκε ήδη είναι τα σύνορα τη ελλάδα με την τουρκία έχουμε ανάγκη την αλληλεγγύη τη ευρώπη υπόθηκε ήδη του πόρου την τεχνογνωσία το ανθρώπινο δυναμικό για να ενισχύσουμε και να φυλάξουμε τα σύνορά μα πιο αποτελεσματικά. ταυτόχρονα όμω είναι και επιτακτική ανάγκη να απαιτήσουμε από την τουρκία να σταματήσει επιτέλου να δίνει τέτοια προκλητική ανοχή στα κυκλώματα και του διακινητέ που εκμεταλλεύονται και την απουσία θεωρήσεων στα σύνορα τη τουρκία με πολλέ γειτονικέ τη χώρε και βεβαίω να δέχεται πίσω του παράνομου μετανάστε που προωθούνται στην ευρώπη μέσα από το έδαφο τη. να ολοκληρωθεί επιτέλου η συμφωνία για την επανεισδοχή όσου ζητούν διεθνή προστασία αναφέρθηκε ήδη α προχωρήσουμε σε μια δικαιότερη κατανομή ευθυνών για την εξέταση των αιτημάτων του και αναφέρομαι προφανώ στην αλλαγή του δουβλίνου 2. αν μου πείτε ότι και σε άλλα κράτη μέλη κύριοι συνάδελφοι υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα θα σα απαντήσω ότι κάνετε λάθο. στι χώρε σα δεν εισέρχονται καθημερινά περίπου 400 μετανάστε. θα σα δώσω λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε λίγο πιο αργά διότι δεν σα προλαβαίνουν οι διερμηνεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε στις χώρες σας κύριοι συνάδελφοι δεν εισέρχονται καθημερινά 400 περίπου παράνομοι μετανάστες με βάση μόνο τα στοιχεία της Frontex και μόνο με τις συλλήψεις. Η πραγματικότητα δηλαδή είναι ακόμη μεγαλύτερα νούμερα. Στη χώρα σας σίγουρα δεν ανεβαίνει καθημερινά στις δημοσκοπήσεις γιατί έχουμε και προεκλογική περίοδο ένα ακροδεξιό κόμμα που προτείνει να μπουν νάρκες με ακούτε νάρκες κατά μήκος των χερσαίων μας συνόρων με την τουρκία ή δεν ξέρω αν συχνά ακούτε προτάσεις της χώρας σας του τύπου να γενικευθεί το δικαίωμα των ιδιωτών στην οπλοφορία. η ευρώπη καθυστέρησε δραματικά να πάρει αποφάσεις και να λάβει μέτρα για την κρίση χρέους στην ελλάδα. Σας... ας μην επαναλάβει το ίδιο σφάλμα στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Η κυρία Μποσκούρ, για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ε, αξιότιμη Πρόεδρε και Επίτροπε, Φαίνεται ότι η Ελλάδα πρόκειται να κλείσει σε ε, στρατόπεδα ε, τους μετανάστες, είτε έχουν ζητήσει άτσιλο είτε όχι, γιατί θεωρεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Ότι είναι, λέει, άρρωστοι ή ζουν σε εκτρές συνθήκες, κέντρα κράτησης, επιχειρήσεις σκούπα από τα κέντρα των πόλεων, ε, τάσεις ρατσιστικές και ξενόφοβες αυξάνονται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν ε, τηρεί τις υποχρεώσεις της ε, ε, σε σχέση με πολίτες τρίτων χωρών. Αυτοί ζουν στη φτώχεια και εσείς τους βοηθάτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς. Τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται για να κλείνονται σε κέντρα κράτησης αυτοί οι άνθρωποι. Δεν καταπολεμάται η ξενοφοβία και ε, ο εξτρεμισμό. Είναι δύσκολη οικονομική καιρή και θα πρέπει εκεί να δοθεί προσοχή. και ολοκληρώθηκε ο κύκλος ε, των εγγεγραμμένων ομιλητών. Θα περάσουμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπασέσκου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με ελληνικά στατιστικά στοιχεία, Το 90% των μεταναστών που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 ήρθαν διαμέσου τη Ελλάδο. Οποιαδήποτε χώρα θα είχε τεράστιε δυσκολίε αν αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συνεκτική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θέλουμε να διαγυριστούμε τέτοιε περιπτώσει. Και όλε οι γείτονε χώρε θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα των μεταναστευτικών ωρεών και τη διασφάλιση των συνόρων. Η Frontex διαδραματίζει σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειές της ε, και να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές οι μετανάστες θα πρέπει να λαμβάνουν γρηγορότερα ε, νόμιμη άδεια παρανομονής και οι διαδικασίες διεκπαιρέωσης των αιτήσεων ασύλου θα πρέπει να επιταχυνθούν. Εχθές η, η Ελλάδα ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα επαναπατρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, διότι ε, ε συμμετέχουν και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα πρέπει να ειδωθεί ως μια ανθρωπιστική κρίση, όπου όλοι μαζί ως ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να δώσουμε μια ενιαία λύση. η χώρα μου δέχεται ετησίως πάνω από 150.000 παράτυπους μετανάστες ποσοστό που πλησιάζει το 15% του συνολικού πληθυσμού της χώρας κάθε χρόνο. οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να γλιτώσουν από τις διώξεις τον πόλεμο και την πείνα και αναμφίβολα δικαιούνται ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης όμως η ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί μόνη της να διαχειριστεί μεταναστευτικές ροές τέτοιου μεγέθους γιατί όπως πολλοί ομιλητές επισήμαναν η ελλάδα υποδέχεται σχεδόν το 90 των μεταναστών που επιχειρούν να μπουν στην ευρωπαϊκή ένωση και το δουβλίνο 2 τους εγκλωβίζει στη χώρα φυσικά τα προβλήματα στην υποδοχή και φύλαξη των παράτυπων μεταναστών είναι μεγάλα και φυσικά η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου παρά τις βελτιώσεις δεν είναι όσο σύντομη θα έπρεπε να είναι. είναι όμως υποκριτικό να συγκρίνεται η ελλάδα με άλλες χώρες της ένωσης στους όρους υποδοχής στη διαδικασία χορήγησης ασύλου δεδομένου ότι το πρόβλημα δεν έχει καμία σύγκριση το μεταναστευτικό ζήτημα στην ελλάδα θα βρει απάντηση μόνο αν αντιμετωπιστεί όπως πραγματικά είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που χρειάζεται πανευρωπαϊκές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα επίση και θα πρέπει να λυθεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράδειγμα με την αναμόρφωση του Δουβλίνου 2 και με ε, ε, επενδύσεις στο ελληνικό σύστημα ασύλου. Αλλά τα χρήματα θα δαπανηθούν στην Ελλάδα. Εκεί είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία εκδηλώνονται και στην υλοποίηση και στην έκθεση ε, του Εθνικού Σχεδίου της Ελλάδας. Η νέα υπηρεσία ασύλου από 700 θέσεις που έχει οργανόγραμμα ε, έχει προσλάβει μόνο 11 άτομα και ε, μόλις άνοιξε και λειτουργεί το Σάββατο πρωί. Δεν βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Επίσης στα κέντρα κράτησης έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες γιατί είναι λιγότεροι οι κρατούμενοι. Μα γιατί δεν θέλει κανείς να κρατά ανθρώπους που ζητούν άσυλο. Βεβαίω είναι πολλά τα προβλήματα και δεν βοηθάει τώρα στην προεκλογική εκστρατεία να χρησιμοποιούν οι μετανάστες ε, ως εκλογικό ζήτημα. Αυτό αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους μετανάστες θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να ζήσουν αξιοπρεπώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καθένας στο μερίδιό του, όχι μόνο οι Έλληνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω στη συζήτηση μερικά πράγματα. Από τη μια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να βάλει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, υπό την ε, κυδαιμονία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ε, καταργεί το Δουβλίνο 2 και από την άλλη μας λέτε ότι είναι σημαντικό το Δουβλίνο 2 για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αντίφαση. Είναι ανοιχτά τα σύνορα, ξέφραγο αμπέλι ακούμε, η Τουρκία δεν βοηθάει, δεν συνεργάζεται, ε, και ε, όσα προγράμματα οικονομικά και αν έχουμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ειλικρινά και να παραδεχθούμε ότι και ο φράχτης δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά τουλάχιστον ένα πρώτο μέτρο. Γιατί συχνά ξεχνάμε και τον πληθυσμό των περιοχών εκεί. Έχει δικαίωμα ο, ο πληθυσμός εκεί, οι Έλληνες, να, να ακουστεί η φωνή τους και να προστατεύονται. Πολύ και τελευταίος ομιλητής στη διαδικασία του Κάτσου Διάε, ο κύριος Γιακολίνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται ένα χρόνο μετά από μια άλλη συζήτηση η οποία στην ουσία είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Πριν από ένα χρόνο, όπως και φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χώρες ε, επιτέθηκαν όλοι στη Λαμπεντούζα. Τώρα στην Ελλάδα το είπε μόλις και ο κύριος Μπουσουτήλ. 60.000 άτομα κατέφτασαν στη Λαμπεντούζα αλλά φυσικά δεν ήθελαν να μείνουν στη Λαμπεντούζα. Αυτοί οι οικονομικοί μετανάστε φτάνουν στην Ιταλία, όπω φτάνουν και στην Ελλάδα, όπω φτάνουν και στη Μάλτα, όχι για να μείνουν ε, σε αυτή την πραγματικότητα. Θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Επομένω, η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη. Η απάντηση είναι μεγαλύτερη ευθύνη, μεγαλύτερη ε, διαχείριση, σωστότερη διαχείριση. Θα ήθελα να προτείνω στην Επίτροπο που έχει ανοιχτή διαπραγμάτευση για τους πόρους που αφορούν αυτό το τομέα παρέμβασης για το διάστημα 2014-2020 θα πρέπει να φροντίσει να κάνει καλύτερες παρεμβάσεις και να εξετάσει καλύτερα τα θέματα. Το ίδιο προτείνω και στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να υπερκεράσουμε αυτό το πρόβλημα διότι η Ευρώπη υπ' αυτό το πρίσμα δεν πάει πουθενά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακολίνο, Επίτροπος μας. Με ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι άκρος ε, σημαντική και δεν αμφιβάλλω ότι θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει πηγόντως μερικά πράγματα. Θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται στο πρόγραμμα δράσης για να δημιουργηθούν σωστές συνθήκες σε κέντρα υποδοχής για να ελέγχεται ο κόσμος να καταγράφεται και να δίνεται συνέχεια στις αιτήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που είναι αυτό τον καιρό στην περιοχή του Εύρου και βρίσκονται σε πολύ εκτρή κατάσταση, ιδιαίτερα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες. Επίσης ε, χρειάζεται να προστατεύονται καλύτερα τα σύνορα και ένα σύστημα επαναπρόθεσης μετά από τις σωστές διαδικασίες όταν θεωρείται ότι δεν χρειάζονται διεθνή προστασία. Και επίσης να αναμορφωθεί η διοίκηση έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ε, τα κονδύλια με σωστό τρόπο. Είναι ε, πάρα πολλά τα λεφτά, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα πρέπει να τα απορροφούν οι ελληνικές αρχές, να είναι σε θέση να το κάνουν. Είμαι πεπισμένη ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα για να ε, επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να σπάσει η γραφειοκρατία. Έχουν γίνει πρόοδοι παντού, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότεροι. Και σε όλες τις διαδικασίες θα συνεχίζουμε να βοηθούμε την Ελλάδα και με χρήματα και ε, το Γραφείο για το Άσυλο είναι εκεί πρόθυμο να συνεργαστεί χέρι με χέρι με τις ελληνικές αρχές. Και επίσης το πρόγραμμα δράσης που αναφέρατε, τη στελέχωση, είναι πραγματικά οξύτατο πρόβλημα. Είναι επιτόπου η Frontex, η Europol για να αντιμετωπιστούν θέματα τράφικινγκ, εμπορίας ανθρώπων, εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικές οργανώσεις για να βοηθήσουν. Το Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης η αρμοστία για τους πρόσφυγες και άλλοι. Και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Ελλάδα στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, να αναλάβει περισσότερες ευθύνες η Τουρκία. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την Τουρκία στη διοικητική της μεταρρύθμιση και οικονομικά για να μπορέσουν και εκείνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, το μερίδιο που τους συναλλογεί. Γίνεται πρόοδος είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Ουδής αμφισβητεί τις τεράστιες δυσκολίες που ε, ζει σήμερα η Ελλάδα. Η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί κόσμος υποφέρει σήμερα στην Ελλάδα και το ξέρουμε. Έχουμε επίγνωση. Επίσης γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε μεταναστευτικές ροές. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και πολλοί θα ε, ζητήσουν να περάσουν από την Ελλάδα για να έρθουν ε, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ευρωπαϊκό το θέμα, το μέλημα και ανησυχία. Θα συνεχίζουμε να βοηθούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο, χέρι με χέρι. Ουδή αναμένει να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη αλλαγέ. Θα χρειαστεί χρόνο. Αλλά θα πρέπει να γίνεται συνεχή διαρκή πρόοδο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συνεργασία των ε, ηθινόντων για να ε, ελέγχουν όλα οι ελληνικές αρχές. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, για την υποστήριξη, για την κατανόησή σας και κυρία Πρόεδρε είμαι βέβαια ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε Επίτροπε Μάλστρομ, τώρα εκ του Συμβουλίου, ο Υπουργό Πέτσικοφ Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι το λόγο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα φλέγων για όλους μας. Η κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την μετανάστευση είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε, να δούμε προσεκτικά τι προκλήσεις αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε σχέση με τη μετανάστευση. Όπως σωστά είπε η Επίτροπος Μάλστρομ, Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα απαιτεί πολλή δουλειά για να αντιμετωπιστεί. Πρέπει και εμείς να δουλέψουμε όμως μαζί με τους Έλληνες. Πρέπει να αποδείξουμε την αλληλεγγύη μας. Υπάρχει σοβαρή μεταναστευτική πίεση. Και πρέπει να αλληλοϊποστηριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θα πρέπει η στήριξή μας να είναι τέτοια, ώστε κάθε κράτος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει απροσδόκητες μεταναστευτικές πιέσεις σεβόμενο ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις του ποπορέων από το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν κρίσεις στα συστήματα αντιμετώπισης της μετανάστευσης των κρατών μελών. Και αν στηρίξουμε την Ελλάδα, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αν προκύψει μια τέτοια κρίση, την μεμονωμένη χώρα μπορούμε να τη συνδράμουμε. Αυτό λοιπόν θα πράξουμε και στην περίπτωση της Ελλάδας. Νομίζω παράσχοντας ε, στήριξη κατά αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε πολύ σύντομα σε ένα σύστημα παροχής ασύλου στην Ελλάδα που και αποτελεσματικό θα είναι και ε, θα μπορεί να αντιποκριθεί σε τέτοιες προκλήσεις με τρόπο εύστοχο και σκόπιμο. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τη συνεργασία που προκύπτει από το Δουβλίνο. Σα ευχαριστώ για αυτή την πλούσια συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι απόψει σα ε, και μα διαφωτίσανε για το όλο ζήτημα. Βεβαίω πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή, διότι η πρόκληση είναι τεράστια για την Ελλάδα και στην πραγματικότητα είναι τεράστια πρόκληση για την ευρωπαϊκή συνεργασία. And, uh, thank you Ευχαριστούμε Υπουργέ, ευχαριστώ όλου για μια συζήτηση που τη θεωρώ ιδιαίτερα επικοδομητική. Η συνεδρίαση διακόπτεται και θα επαναληφθεί στις 9 η ώρα ακριβώς.